στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ε, είναι ανάξιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το οποίο συμβαίνει. Τιμωρούμε δηλαδή α, αυτούς που δεν φταίνε. Πρέπει να φύγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Ε, επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η προφορική ερώτηση στην Κομισιόν για την απαλλαγή κατά κατηγορία για μηχανοκίνητα οχήματα. Κύριο Στόγιαν. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων έθεσε αυτό το ερώτημα γιατί έχει υπάρξει μία αναθεώρηση του κανονισμού απαλλαγής ε, των ε, μηχανοκίνητων οχημάτων. Και πρέπει να το δούμε προσεκτικά. Όπως ξέρετε, οι κανονισμοί εξαίρεση είναι πάρα πολύ σημαντικοί για τι επιχειρήσει. Ο κανονισμός αυτός υιοθετήθηκε το 2002. Τότε η Κομισιόν θεώρησε πως υπήρχε ολιγοπόλιο στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτων. Οι έξι μεγαλύτεροι κατασκευαστές ε, στην Ευρώπη είχαν ένα 75% της αγοράς. Με βάση αυτά η Κομισιόν αποφάσισε, θεώρησε πως ο τομέας αυτός δεν θα πρέπει να υπαχθεί στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής κατά κατηγορία και υιοθέτησε συγκεκριμένο κανονισμό. Ο κανονισμός αυτός θα εκπνεύσει την 31η Μαΐου τρέχοντος τώρα, η Κομισιόν θεωρεί πως η αγορά νέων οχημάτων είναι πολύ ανταγωνιστική και πως τα επίπεδα συγκέντρωσης έχουν μειωθεί. Οι συνέπειες, ε, ως συνέπεια αυτής της αξιολόγησης η Κομισιόν ε, προτείνει ε, πως δεν χρειάζεται συγκεκριμένος κανονισμός για την πώληση νέων αυτοκινήτων και εμπορικών οχημάτων. Προτείνει να υιοθετηθεί κανονικό κανονισμό απαλλαγής μόνο για επισκευές και ανταλλακτικά. Μας απασχολεί λοιπόν στο Κοινοβούλιο. Όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια εξαιρετική οικονομική κρίση και τα ποσοστά ανεργία είναι πάρα πολύ υψηλά. Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία είναι ένα κλάδο κλειδί και συνεισφέρει στην απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Πιστεύουμε πως πρέπει να υπάρχουν γενικοί όροι για να γίνει αηφόρος αυτός ο τομέας και να παραμείνει οικονομικά αποτελεσματικός και πράσινος. Επίσης πρέπει να διασφαλίσουμε πως και οι μικρομεσαίες εταιρείε ε, θα έχουν ε, ευνοϊκούς όρους. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε την σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως ε, προμηθευτών θέσεων εργασίας. Όμως πάρα πολλοί αντιπρόσωποι αυτοκινήτων και συνεργεία έχουν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο λέγοντας πως θα οδηγήσει σε περαιτέρω επιδίνωση των σχέσεων ισχύω μεταξύ των κατασκευαστών και της υπόλοιπης αλυσίδας. Γι' αυτό κύριε Αλμούνια, θα ήθελε η Επιτροπή μας να σας ρωτήσει πρώτα απ' όλα ποια αποτελέσματα ανάλυσης αγοράς οδήγησαν την Κομισιόν να συμπεράνει πως η πρωτογενής αγορά είναι αυτή τη στιγμή αποτελεσματική και η αγορά με... η δευτερογενής είναι προβληματική. Δεύτερον, πώς αξιολογεί η Κομισιόν την σχέση ισχύω μεταξύ κατασκευαστών και εμπόρων αυτοκινήτων υπό τον τωρινό κανονισμό και υπό το προτινόμενο πλαίσιο. Θεωρείτε πως είναι απλούστερη η κατάσταση ή υπάρχει μια συλλογική δεσπόζουσα θέση. Τρίτον, πώς σκοπεύει η Κομισιό να παρακολουθήσει την εξέλιξη των σχέσεων αυτών στην πρωτογενή αγορά και στην αγορά after sale. Τι σκέφτεται να κάνει η Κομισιόν θα πρέπει να δούμε πώς τα πράγματα έχουν χειροτερεύσει την πρωτογενή αγορά. Τέταρτον, ποιο είναι ο αναμενόμενο αντίκτυπο του νέου νομοθετικού πλαίσιου στην κατανάλωση, ειδικά στην τιμή και στου όρου που προσφέρονται. Πέμπτον, ποια σχόλια λάβατε από του ενδιαφερόμενου κατά τη διάρκεια τη διαβούλευση και σκοπεύει η Κομισιόν να τα ενσωματώσει στο τελικό νομοθετικό πλαίσιο. Και τέλο, η Κομισιόν συμφωνεί να εξετάσει την εναρμόνιση της νομοθεσίας στον τομέα της διανομής με την αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας έτσι ώστε όλοι οι έμποροι να έχουν το ίδιο επίπεδο συμβατικής προστασίας σε όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Χάρμπορ, ευχαριστώ. Εξ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή χαίρομαι που μπορούμε να προβάλλουμε και το δικό μας ερώτημα και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή που κατέχει ηγετικό ε, ρόλο σε θέματα ανταγωνισμού διότι αυτό είναι ένα θέμα που άπτεται της πολιτικής ανταγωνισμού και είναι ύψης της σημασίας για τους καταναλωτές ορισμένα στοιχεία υπέρ του καταναλωτή εκφράζονται πολύ καλά. Θα ήθελα να πω ότι τα στοιχεία της πρότασης της Κομισιόν που σχετίζονται με τις πωλήσει σέρβις και επισκευή σχετίζονται με τα συμφέροντα των καταναλωτών που δείξαμε στη δική μας Επιτροπή και όχι στα πλαίσια της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, αλλά σε σχέση με πληροφορίες στον τομέα του σέρβις και των επισκευών. Συνεργαστήκαμε και με την Επιτροπή Περιβάλλοντος σε σχέση με προδιαγραφές περιβάλλοντος στα μηχανοκίνητα οχήματα και νομίζω ότι τα στοιχεία που έχουν ενισχυθεί είναι ευπρόσδεκτα σε σχέση με την βιώσιμη ανταγωνιστικότητα ως προς τις επισκευές και αγορές εξαρτημάτων, ανοίγοντας αυτή την αγορά. Η μόνη επιφύλαξη που ε, σε σχέση με το ψήφισμα αφορά τη διαθεσιμότητα πληροφοριών. Δεν είμαστε πεπισμένοι και ίσως θέλετε να σχολιάσετε, δεν είμαστε πεπισμένοι ότι, δεν είμαστε πεπισμένοι ότι οι κατευθυντήρες γραμμές είναι αναγκαίες έτσι ώστε οι τεχνικές αυτές πληροφορίες να είναι διαθέσιμες. Διότι θα είναι δυνατόν για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να διαθέσουν αυτές τις πληροφορίες σε ηλεκτρονικό μορφότυπο αλλά όχι ε, χρησιμοποιώντας το καταλληλολογισμικό. Άρα δεν θα είναι τόσο χρήσιμα αυτά τα στοιχεία για τις επισκευές. Ως προς τις πωλήσει, ακούσαμε εύγλωτα από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων πολλά ζητήματα, αλλά δεν είμαστε τόσο πεπισμένοι. Δεν ξέρω κατά πόσο λάβατε υπόψη τις ανησυχίες των καταναλωτών. Η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή σε μία ακρόαση όπου ακούσαμε από τους αντιπροσώπους ακούσαμε πάρα πολλά και ελέγχθη ότι ο ανταγωνισμός, ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία υπέρ του ανταγωνισμού στην ε, αγορά πωλήσεων, αλλά δεν ανταποκριθήκατε στις ανησυχίες μας. Ε, δηλαδή, δείξατε μεγάλο ζήλο να απλουστεύσετε πράγματα για να κάνετε τη ζωή σας, τη δική σας ζωή ευκολότερη. Ίσως ανακύπτουν προβλήματα από αυτό. Αλλά θα ήθελα να δείτε τα αποδεικτικά στοιχεία της ακρόασης. Δηλαδή, οι αντιπρόσωποι και οι καταναλωτές έχουν μεγάλες ανησυχίες σε σχέση με την διανομή, με το δίκτυο διανομής ως προς τις ε, συλλήβδην εξαιρέσεις. Και το 2002 με βάση το δίκτυο ε, διανομής θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να επανακτήσουμε ένα σωστό πλαίσιο ε, διανομής και κατανομής ως προς τους αντιπροσώπους. Τότε το σύστημα ήταν λειτουργικό. Αν δείτε την αγορά, αυτό ισχύει. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, γιατί τότε δεν ήσασταν παρόν, κύριε Επίτροπε, ότι έγινε υπήρξαν πολύ ισχυρά λόμπι στην αυτοκινητοβιομηχανία. Τώρα τι μας λένε οι αντιπρόσωποι αυτοκινήτων ότι αυτές οι διατάξεις είναι πολύ αδύναμες, ενώ οι κατασκευαστές τις βρίσκουν πολύ καλές. Δεν λέω ότι πρέπει να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία. γιατί πρέπει να εφαρμόσουμε αυτό το πλαίσιο σε λίγες μέρες. Λέμε όμως στο ψήφισμα δείτε τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Και θα ήθελα να σας πω και το εξής. Ο Επίτροπος Μπαρνιέ θα υποβάλει μία έκθεση για τον ανταγωνισμό στην αλυσίδα ε, λιανικής. Τα μηχανοκίνητα θα πρέπει να ενταχθούν εκεί γιατί χρειαζόμαστε μία συνεκτική πολιτική από την Κομισιόν. Και δεύτερον, τα έγγραφα που είδα των υπηρεσιών σας λένε ότι πρόκειται για μία ε, προπαρασκευή για τα νέα πράσινα οχήματα, ηλεκτρικά οχήματα. Διαβάσαμε και το έγγραφο του κυρίου Ταγιάννη. Θα ήθελα τον επόμενο χρόνο να δείτε τα έγγραφα του, του κυρίου, των κυρίων Ταγιάννη και Μπαρνιέ και να μας διασφαλίσετε ότι αυτό είναι το σωστό έτσι ώστε να έχουμε κάποια αξιοπιστία, διότι δεν είμαστε καθόλου πεπισμένοι για τα σχέδιά σας. Ευχαριστούμε κύριε Χάρμπορ. Ο Επίτροπος, ο κύριος Σαλμούνια, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. κανονισμός ε, απαλλαγής κατά κατηγορία για τα αυτοκίνητα εκπνέει την 1η Ιουνίου και πρέπει να υιοθετηθεί άρα ένας νέος κανονισμός. Οπότε η Επιτροπή έθεσε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη 26 Μαΐου. Η πρόταση που συζητάμε τώρα στις υπηρεσίες μας και σε λίγες ημέρες με τα γραφεία μας προετοιμάζοντας ε, μια συνεδρίαση του σώματος βασίζεται σε μια, εμβάθος, σε μια εισβάθος ανάλυση. Ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2006 η δημόσια διαβούλευση. Πέρσι το Δεκέμβρη, μετά από 3,5 χρόνια, δημοσιεύσαμε τα σχέδια κατευθυντηρίων γραμμών. Καθ' όλη τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι, το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη αναμίχθηκαν. Και λάβουν υπόψη πολλά επιχειρήματα. Σε έγιναν πολλές συζητήσεις, εργαστήρια, πρωτοβουλίες, και εδώ μέσα, στο Κοινοβούλιο. Η τελευταία έλαβε χώρα στις 12 Απριλίου φέτος στην Επιτροπή Οικονομικών. Ποια είναι τα κύρια συμπεράσματα αυτής της ε, μακροσκελούς ε, διαβούλευσης. Πρώτα απ' όλα μάθαμε κάτι θετικό, πως ο καταναλωτής στην Ευρώπη απολαμβάνει έντονο ανταγωνισμό. Στην ετήσια έκθεση τιμών αυτοκινήτων εξετάσαμε 80 μοντέλα 25 κατασκευαστών. Οι τιμέ δεν είναι ο μόνος παράγων που μας λένε πω ο ανταγωνισμό λειτουργεί. Υπάρχει μεγαλύτερη επιλογή από ό,τι πριν από 10 χρόνια, περισσότερες μάρκες επίσης για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε πως οποιοδήποτε κατασκευαστής έχει δεσπόζουσα θέση είτε από μόνο του είτε συνεργασία με άλλου. Το τρέχον καθεστώς ε, περιέχει κανόνε ε, που ήταν λογική το 2002 όταν αναμέναμε συγχωνεύσει στον τομέα των αυτοκινήτων. Η περίοδο αυτή δεν συνέβη τελικά και ανταυτού σήμερα έχουμε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά. Με το να επιτρέψουμε περισσότερη ευελιξία για την διανομή οχημάτων θα αποκαταστήσουμε τα κίνητρα των κατασκευαστών για να μειωθεί το κόστος πώλησης αυτοκινήτων. Να υπενθυμίσω πως το κόστος της διανομής κυμαίνεται γύρω στο 30% της τιμής ενός καινούργιου αυτοκινήτου. Με το να μειώσουμε αυτό το κόστος, οι κατασκευαστές ε, θα βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση και θα ωφεληθεί ο καταναλωτής. Γνωρίζω πως υπάρχουν κάποιες ανησυχίες ε, σε σχέση με πωλήσει διαφορετικών μαρκών και συμβατική προστασία των εμπόρων, κάτι το οποίο αναφέρατε και οι δύο. Να τονίσω πως υπάρχει αυτή η πώληση διαφορετικών μαρκών και θα συνεχίσει να υπάρχει εκεί όπου το απαιτεί η πραγματικότητα της αγοράς. Αυτό συμβαίνει σε χώρες με πολύ μεγάλους εμπόρους που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διανομές πολλών εταιριών όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε αραιοκατοικημένες περιοχές όπου είναι λογικό να πουλάνε διάφορες μάρκες οι ε, πολιτές. Αυτό συνέβαινε και στο παρελθόν πριν το 2002 και παραμένει πραγματικότητα 8 χρόνια μετά. Αλλά ο κανόνας τότε και τώρα είναι μία μάρκα. Αυτό το οποίο παρατηρήσαμε είναι πως οι κατασκευαστές καταφεύγουν σε άλλες μορφές ε, διανομής, μεταξύ των οποίων και δικά τους καταστήματα. Το τι γίνεται στη Γερμανία, παραδείγματο χάρη, είναι χαρακτηριστικό. Καθώς 67% των αυτοκινήτων πολλούνται μέσω δικτύων εμπόρων και αυτό ήταν 90% πριν το κανονισμό του 2002. Παρ' όλα αυτά, Απαντήσαμε στις ανησυχίες που εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένης και τη διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και έχουν εισαχθεί εδώ πέρα κάποιες δικλείδες ασφαλείας για αντιπροσωπείες με πολλές μάρκες. Προτείνουμε μια μεταβατική φάση λοιπόν κατά τη διάρκεια της οποίας θα εφαρμοστεί ο τρέχον κανονισμός μέχρι το τέλος του 2013 για να υπάρχει αρκετός χρόνος σε όσους έχουν επενδύσει σε πολλές μάρκες να αποσβέσουν την επένδυσή του. Γιατί σκοπεύουμε τώρα να καταργήσουμε αυτές τις ρήτρε που προστατεύουν συμβατικά τους ε, εμπόρους. Γιατί δεν είναι το δίκαιο του ανταγωνισμού το κατάλληλο για να δούμε την ανισορροπία δυνάμεων μεταξύ των συμβαλωμένων μερών. Τα ζητήματα αυτά ανήκουν στη σφαίρα του εμπορικού δικαίου σε μια ανταγωνιστική αγορά όπως η αγορά του αυτοκινήτου ο... το δίκαιο του ανταγωνισμού δεν θα πρέπει να επισέρχεται στην ισχύ των συμβαλωμένων μερών καθώς κάτι τέτοιο θα αποτελούσε παρέμβαση και πρέπει να είμαστε αναλογικοί στις παρεμβάσεις μας. Στην διαβούλευση επίσης μάθαμε και κάποια άλλα πράγματα, ίσως όχι τόσο θετικά. Σε αντίθεση με τις τιμές των αυτοκινήτων, η τιμή της επισκευής αυξήθηκε. Οι επισκευές και η συντήρηση είναι πολύ σημαντικές για τους καταναλωτές, όχι μόνο για λόγους ασφάλειας και αξιοπιστίας, αλλά και γιατί αυτές αποτελούν το 40% της αξίας α, ιδιοκτησίας ενός αυτοκινήτου. Και βεβαίως εμποδίζονται ακόμα τα ανεξάρτητα συνεργεία να ανταγωνιστούν καθώς ε, έχουν μειωμένη πρόσβαση σε ανταλλακτικά και τεχνικές πληροφορίες. Οπότε η μεταρρυθμισή μας σκοπεύει να επιτρέψει στα ανεξάρτητα συνεργεία να έχουν καλύτερη πρόσβαση και να μην αποκλείονται από την αγορά από άλλες νέες πρακτικές. Έτσι θα έχουμε καλύτερη ποιότητα και χαμηλότερες τιμές. Καταλήγοντα, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω πως το νέο πλαίσιο θα είναι καλύτερο για τους καταναλωτές. Η βασική μας προτεραιότητα είναι να αυξηθεί ο ανταγωνισμός στην αγορά μετά την πώληση. Παρά το ότι οι κατασκευαστέ μπορεί να έχουν ισχυρή εμπορική θέση έναντι των εμπόρων, ανταγωνίζονται μεταξύ τους και σήμερα δεν υπάρχει λόγο να αποκλίνουμε και να διατηρηθεί ο ανταγωνισμός σε αυτές τις συμφωνίες από τον κανονισμό απαλλαγή που υιοθέτησε πρόσφατα η Κομισιόν και ο οποίο επίση θα τεθεί ενισχύ στο τέλο του μήνα. Πράγματι, η Κομισιόν και συγκεκριμένα η δική μου Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού θα παρακολουθήσει στην τομέα προσεκτικά και δεν πρέπει να έχουμε αμφιβολία για την αποφασιστικότητα της Κομισιόν να εφαρμόσει τους κανόνες και να κάνει τα απαραίτητα βήματα εάν διαπιστώσουμε τυχόν παραβιάσεις. Περνάμε στους ομιλητές εξ ονόματος των ομάδων. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Κάρας. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε πολλά. Με την προφορική αυτή ερώτηση και το ψήφισμα θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους εμπόρους αυτοκινήτων, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν μια φωνή, να ακουστεί η φωνή τους. Γιατί αυτή τη φωνή δεν την άκουσε η Κομισιόν τα τελευταία χρόνια. Στις ακροάσεις ακούστηκαν αμφιβολίες περί άνησης μεταχείρισης των εμπόρων από τους κατασκευαστές. Μιλήσαμε για νομική ανασφάλεια έγινε λόγος για μείωση του ανταγωνισμού μέσω των προβλημάτων που έχουν οι μικρομισές ε, αυτές επιχειρήσεις, αλλά δεν λάβαμε απάντηση. Σας απευθύνω έκκληση στο 12 παρά 1. Να εκμεταλλευτείτε τις 21 ημέρες μέχρι τις 26 Μαΐου για να ενσωματώσετε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου στον κανονισμό σας να έρθετε πιο κοντά στους εμπόρους αυτοκινήτων χωρίς να αλλάξει την γενικότερη κατεύθυνση της Κομισιόν. Ακούστε το Κοινοβούλιο, πάρτε σοβαρά τους εμπόρους αυτοκινήτων και βοηθήστε τις μικρομεσαίες αυτές τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Για μισή λεπτό έχει το λόγο ο κύριος Λούντβικσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω τέσσερα υποζητήματα σε αυτή τη συζήτηση. Είναι ατυχές το γεγονός ότι οι μικρές και μεγάλες εταιρείες αλληλοανταγωνίζονται. Θα πρέπει να ορίσουμε ένα πλαίσιο στο οποίο να μπορέσουν να συνεργαστούν. Δεύτερον, είναι πολύ θετικό οι βελτιώσεις στον τομέα της ανταγωνιστικότητας προς, ως προς τις νέες πωλήσει αυτοκινήτων. Τίποτα δεν είναι αδύνατον λοιπόν. Άρα μακροχρόνια θεωρούμε ότι μπορούμε να τονώσουμε τον ανταγωνισμό. Τρίτον, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθήσει τι συμβαίνει σε σχέση με τα νέα οχήματα και τον ανταγωνισμό. Θα πρέπει να δοθούν, να υπάρξουν μέτρα συνέχειας. Όλοι οι τομείς βιομηχανίας θα πρέπει να γνωρίζουν τι θα ισχύει από τον Ιούνιο του 2013. Θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε συζητήσεις για τη μετάβαση στα πράσινα αυτοκίνητα τα οποία δεν μολυνούν τόσο. Οι κανόνες ανταγωνισμού θα πρέπει να είναι ευέλικτοι σε σχέση με τις επιδοτήσεις έτσι ώστε να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για την αγορά και επίσης τα οχήματα του περιβάλλοντος να, μην αποτελέσουν πρόσκομα στον ε, τομέα ελιανικής. Ο κύριος Μπουσόη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, πιστεύω ότι ε, έχει μεγάλη σημασία η ύπαρξη μηχανοκίνητων για τους μικρούς καταναλωτές, έτσι ώστε να μπορέσουν οι μικροί καταναλωτές να αγοράζουν οχήματα χωρίς να καταβάλουν ένα πολύ υψηλό κόστος. Γι' αυτό ανησυχώ για τις μαζικές εξαιρέσεις και τις επιπτώσεις για τους καταναλωτές. Άκουσα τα επιχειρήματα του ε, Επιτρόπου. Μας τόνισε για το γεγονός ότι οι στόχοι έχουν επιτευχθεί και υπάρχει επαρκές επίπεδο ανταγωνισμού. Δεν τάσσομαι υπέρ της άρσης των ε, ε, μαζικών αυτών εξαιρέσεων. Θα πρέπει όμως σε μια μεταβατική φάση να κρίνουμε κατά πόσο ισχύει αυτή η υπεροχή και η δεσπόζουσα θέση ορισμένων βιομηχανιών αυτοκινήτου. Θα ήθελα να είμαι σίγουρος ότι δεν θα υπάρξει δεσπόζουσα θέση ως προς το μέρισμα της αγοράς για τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες. Επίσης, η μαζική αυτή εξαίρεση δεν θα πρέπει να ισχύσει και στον τομέα των εξαρτημάτων και των επισκευών σε σχέση με τις πωλήσει. Νομίζω ότι ότι οι ανεξάρτητες επισκευές γίνονται από εκείνους που τις κάνουν καταχρηστικά και δεν έχουν τις κατάλληλες πληροφορίες. Άρα περιορίζονται οι καταναλωτές και ελπίζω η Επιτροπή να αλλάξει αυτό το πλαίσιο. Θα ήθελα λοιπόν η Επιτροπή να μας πει ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για να αποφευχθούν καταστάσεις που είναι επώδυνες για τον καταναλωτή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Μπουσόη. Ο κύριος Σιμάνσκι για ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε πως τα ανταλλακτικά κατά 80% προέρχονται από ανεξάρτητους κατασκευαστές. Έχουν όμως τεράστιο πλεονέκτημα οι κατασκευαστές και εναντί των ανεξάρτητων συνεργείων και των ανεξάρτητων κατασκευαστών. Δεν πρέπει λοιπόν να είναι ολιγοπολιακή η κατάσταση. Πρέπει να εγγυηθούμε στους ε, πολίτες μας την ελεύθερη επιλογή συνεργείων και ανταλλακτικών και, και πληροφόρηση. Επίσης να δούμε και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία τα οποία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν και εργαλεία και ανταλλακτικά από ανεξάρτητους προμηθευτές. Ε, αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες εγγυήσεις όμως θα παραμείνουν όλα αυτά φαντασία μόνο. Και πρόκειται για ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Σας ευχαριστώ. Πάμε στο γύρο των υπολείπων ομιλητών. Ο κύριος Λάγκε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από πλευράς Επιτροπής Βιομηχανίας ακριβώς θέλουμε να προστατεύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο ανταγωνισμός δεν είναι αυτός σκοπός. Αν δούμε την κατάσταση με τους μικρούς εμπόρους και τα μικρά συνεργεία, πρέπει αυτοί να ενισχυθούν όσον αφορά την οικονομική τους δύναμη. θα έχουμε μόνο μεγαλεμπόρους και εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Οπότε θα πρέπει να επιτραπεί η πώληση πολλών μαρκών, θα πρέπει τα συνεργεία και οι έμποροι να έχουν απεριόριστες πληροφορίες για την επισκευή των οχημάτων. Τρίτον, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης προσόντων, ειδικά τώρα που μιλάμε και για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για τη συντήρησή τους δηλαδή και ασφάλεια στην επένδυση. Να μην υπάρχει δηλαδή άλλη αναθεώρηση και προστασία των συμβάσεων. Πρέπει δηλαδή να μπορούν να κάνουν απόσβεση αυτοί οι άνθρωποι στην επένδυσή τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για δύο λεπτά. Ο κύριος Έγγελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να μιλήσουμε για την πραγματικότητα των πολιτών αυτοκινήτων. Στη χώρα μου είναι έντονη η δυσαναλογία μεταξύ των αντιπροσώπων αυτοκινήτων και των αυτοβιομηχανιών ως προς τις απαιτήσει που επιβάλλει αυτή η κινητοβιομηχανία στους αντιπροσώπους. Εδώ δεν παίζει κύριε Επίτροπε ο ανταγωνισμός. Διότι ο ανταγωνισμός είναι μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών και όχι μεταξύ αυτο, αυτοκινητοβιομηχανιών και αντιπροσώπων αυτοκινήτων ε, τι δουλειά έχει το γκαράζ της γωνίας να παρακολεί τον ανταγωνισμό. Το πρόβλημα είναι σε άλλα επίπεδα και αυτή είναι η πραγματικότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μικροί λοιπόν τι ζητάνε από την Κομισιόν. Μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Είναι ο Δαβίδ ενάντια στο Γολιάθι. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες απαιτούν όλο και περισσότερα πράγματα από τους αντιπροσώπους αυτοκινήτων. Είναι λανθασμένα τα επιχειρήματα για την κατάργηση του κανονισμού. Εμείς δεν διαμορφώνουμε καλύτερα την εσωτερική αγορά περιορίζοντας την ελευθερία των αντιπροσώπων. Η κυρία Τικάου, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Το κινητό η αγορά αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβάνει τι συμπεριλαμβάνει την αυτοκινητοβιομηχανία, τους αντιπροσώπους, ε, τους εμπόρους ανταλλακτικών. Υπάρχει πρόβλημα με το εμπόριο ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Θέλουμε η Κομισιόν να κάνει μία διαβούλευση για το θέμα των ανταλλακτικών τα οποία είναι ακριβά και πρέπει να πουλούνται σε ανταγωνιστικές τιμές. Το νέο πλαίσιο θα πρέπει να εγγυάται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ευνοϊκούς όρους και αυτές οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να εξαρτώνται από τους μεγάλους παραγωγούς οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να διευρυνθούν και να λαμβάνουν υπόψη και τον τελικό καταναλωτή. Ευχαριστώ κυρία Τικάου, η κυρία Σάγια. Ε, Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. με αυτά τα οποία ακούστηκαν είναι σαφές πως ε, το Κοινοβούλιο ενισχύει πάρα πολύ ειδικά για τους εμπόρους και για την ισορροπία μεταξύ των ε, κατασκευαστών και βεβαίως για τις υπηρεσίες ε, του χρήστη οδηγού. η ανάγκη αυτής της ισορροπίας καθίσταται σαφής στην Φιλανδία και στις άλλες σκανδιναβικές χώρες όπου πάρα πολλές περιοχές είναι αραιοκατοικημένες. Άρα χρειαζόμαστε ξεκάθαρες προϋποθέσεις έτσι ώστε να έχουμε εγγύηση καλών υπηρεσιών για τον καταναλωτή η αγορά αυτοκινήτων στην Φιλανδία φέτος θα φτάσει τα 100.000 κομμάτια για 5 εκατομμύρια πληθυσμό συνολικά. Οπότε είναι απολύτως απαραίτητο να μην επιδεινωθεί η κατάσταση μέσω αυτών των αλλαγών. Ο κανονισμός μέχρι τώρα αποδείχθηκε καλός και το ερώτημα είναι γιατί να αλλάξει αυτή τη στιγμή. Επίσης η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε καταναλωτές σε αριοκατοικημένες περιοχές δεν θα πρέπει να περιοριστεί. και ειδικά αυτές τις περιοχές πρέπει να τις σκεφτούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Ευχαριστώ. Να δύο λεπτά ο κύριος Κάρας. Κύριε Επίτροπε, μας ακούσατε. Και θέλω να πω πως αυτή είναι η διαφορά μεταξύ θεωρίας και πράξης. Επευθύνω λοιπόν πάλι έκκληση Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είχα πει στον πρόεδρο της Κομισιόν άνοιξη του 2009. Έχουμε αναπάντητα ερωτήματα για τους εμπόρους, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είμαστε μέσω μιας κρίσης και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Η αγορά απασχόλησης είναι βέβαιη. Καλό είναι να παραταθεί ο υπάρχον κανονισμός και όχι να δημιουργηθεί ένας νέος που θα επιτείνει αυτά τα προβλήματα. εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικοί εθνικοί κανονισμοί. Υπάρχει επίσης ένας μη δεσμευτικός κανονισμός, θέλουμε να εφαρμοστεί αποτελεσματικά. Επίσης να υπάρξει μεγαλύτερη ελευθερία για τους εξιοδοτημένους αντιπροσώπους. Επίσης να υπάρχει εγγύηση παροχής πληροφοριών στα συνεργεία. Κάποια πράγματα εντωμεταξύ μένουν απ' έξω όσον αφορά παραδείγματο χάρη τι προθεσμίε καταγγελία συμβάσεων, μεταφορά επιχειρήσεων και την επίλυση διαφορών. Οπότε σας παρακαλώ σκεφτείτε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, χρειαζόμαστε περισσότερο ανταγωνισμό αλλά αυτό δεν θα γίνει με την μείωση των δυνατοτήτων των εμπόρων. Δείτε λοιπόν σοβαρά την αγορά, τις επιχειρήσεις, το ψήφισμα του Κοινοβουλίου και χρησιμοποιήστε τις 21 μέρες που έχετε ακόμα στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ. Πάμε στο Catch the Eye. Για ένα λεπτό. Ο κύριος Ρούμπιχ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Όλοι οι ομιλητές μίλησαν και είναι υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρέπει να υπάρχουν οι μικροί έμποροι που απασχολούν ανθρώπους. Για αυτούς είναι σημαντικό να έχει ανταγωνισμό το σύστημα το ίδιο και για τους ε, εμπορούσα ανεξαρτήτως αν είναι μεγάλη ή μικρή. Ειδικά λοιπόν στον τομέα του αυτοκινήτου μπορεί, πρέπει να έχει και ο καταναλωτής ένα ανταγωνισμό που θα λειτουργεί και όχι ένα μονόμερο, μονομερές σύστημα που δεν έχει πλέον δυνατότητα επιλογής και ακριβώς η δυνατότητα αυτή επιλογής θα αποδειχθεί σημαντική για την ύπεθρο, δηλαδή να υπάρχει συνολική κάλυψη της υπαίθρου. Γι' αυτό θεωρώ πως έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Κάρας όταν λέει πως δεν έχουμε ακόμα πάρα πολύ χρόνο και πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρούμπιχ. Κέλλη. Πρώτα απ' όλα συμφωνούν όλοι πως το αυτοκίνητο δεν είναι πλέον πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Και αυτό κατέστησε σαφέ πριν από δύο εβδομάδε όταν είχαμε την Χριστιακή στάχτη. Και ξαφνικά πλοία, τρένα και αυτοκίνητα χρησιμοποιήθηκαν και εγώ ήμουν στο αυτοκίνητό μου και ποτέ δεν είχα αισθανθεί τόσο ανεξάρτητο. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε του καταναλωτέ να έχουν επιλογέ. αλλά όχι ει βάρο των μικρομεσαίων εμπόρων. Περισσότερε από αυτέ οι επιχείρησει είναι οικογενειακέ σε μικρέ πόλει που προσπαθούν να κάνουν καλές προσφορές, να ικανοποιήσουν την αγορά και έχουν πολλές δύσκολες συνθήκες ανταγωνισμού. Οπότε συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κάρας και η Λυπή πως πρέπει να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα αυτών των επιχειρήσεων στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Úvodom že rozumiem o autoservisu. Σας ευχαριστώ οι προσπάθειες διασφάλισης ελεύθερης επιλογής των καταναλωτών όσον αφορά τα συνεργεία είναι κατανοητές, αλλά υπάρχουν και όρια στην απόρριτη ελευθερία σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή θα σκεφτείτε μια παρομοίωση. Θα μπορούμε να στείλουμε ένα Airbus για service στη Ρωσία. Έτσι δεν μπορούμε να έχουμε και συνεργεία ε, τα οποία δεν θα ακολουθούν τις μεθόδους ε, των ε, κατασκευαστών. Ο πελάτης έχει την ελεύθερη επιλογή αλλά χρειάζεται να μπορεί να αποφασίσει να στραφεί σε ένα συνεργείο το οποίο δεν θα του δώσει πληροφορίε. Εκεί πέρα όμως διατρέχει τον κίνδυνο να μην είναι καλή η επισκευή του αυτοκινήτου. Δεν μπορούμε να αναμένουμε πως όλα τα συνεργεία θα παρέχουν τις ε, ίδιες ε, υπηρεσίες. Εγώ ως καταναλωτής προτιμώ ένα καλό συνεργείο το που έχω μια καλή σχέση μεταξύ εμπόρου και υπάρχει και καλή σχέση βεβαίως μεταξύ εμπόρου και κατασκευαστή και αυτό ωφελεί και τον καταναλωτή. Ο κύριος Αλμούνια. Θέλω να ε, ευχαριστήσω όχι μόνο εσάς για την καταπληκτική σας προεδρία αλλά και για όλους τους βουλευτές ε, και βουλευτίνες για τις τοποθετήσεις τους. Τους ευχαριστώ όχι μόνο για τις σημερινές τοποθετήσεις αλλά για όλες γενικώ τις συνεισφορές τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης προς όλες τις κατευθύνσεις όχι μόνο με το Κοινοβούλιο τα μέλη και τις επιτροπές ε, που ασχολούνται με θέματα ανταγωνισμού, ε, αυτοκινήτων, ε, καταναλωτών κλπ. Αλλά και με τα κράτη-μέλη και όλους τους ενδιαφερόμενους κλάδους και εκείνους που θέλησαν απλώς να πούν τη γνώμη τους. Τα θέματα ανταγωνισμού είναι και στόχος δηλαδή της πολιτικής ανταγωνισμού είναι το πώς θα ευνοηθεί ο καταναλωτής και στόχος δηλαδή της, ε, των ε, ρυθμίσεών μας. Οι καταναλωτές ε, όταν πάνε σε ένα γκαράζ διότι όπως είπατε όλοι αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο κομμάτι του οικογενειακού προπολογισμού. Πάνε λοιπόν στον καράζ και θέλουν να συγκρίνουν τις τιμές και τώρα θα γίνεται αυτό καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Θέλουν να επιλέγουν χωρίς εμπόδια παρακόλλησης του ανταγωνισμού Δηλαδή τώρα η επιλογή τους θα, μεγαλώ, θα αυξηθεί και θέλουν επίσης να επιλέγουν και τα συνεργεία που θα πηγαίνουν το αυτοκίνητό τους. Άσχετα αν αυτά τα συνεργεία είναι συνδεδεμένα ή όχι με τον κατασκευαστή και να έχουν φυσικά αυτά τα συνεργεία και το, την απαραίτητη γνώση και τα απαραίτητα ανταλλακτικά. Όλα αυτά βελτιώνονται με την τωρινή πρόταση της Κομισιόν. Σας παρακαλώ προσέξτε αυτό το οποίο λέει το κείμενο και αυτό που έχετε και τις κατευθυντήριες γραμμές. Θα μας επιτρέψει λοιπόν αυτό το κείμενο να έχουμε καλύτερες συνθήκες. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τι μας πρότειναν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί εμεί ακούμε τις γνώμες όλων. Τι έγινε λοιπόν με αυτούς. Αυξήθηκαν ή μειώθηκαν. Ευνοήθηκαν στο να μπουν δηλαδή στην αγορά της διανομής ή περιορίστηκαν. Το δεύτερο συνέβη. Και δεν ήταν αυτή η βούληση του νομοθέτη το 2002. Αυτό όμως μας το δείχνει η εμπειρία των τελευταίων ετών και αυτό θέλουμε να διορθώσουμε. Τι συμβαίνει μέχρι σήμερα σε συγκεκριμένα, με συγκεκριμένα συνεργεία ή με κατασκευαστές ανταλλακτικών αυτοκινήτων έχουν δυσκολίες να ανταποκριθούν και θα, εξαφανιστούν. Εμείς θέλουμε να τους δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες στις ΜΜΕ σε όλη την αλυσίδα, δηλαδή από την κατασκευή των ανταλλακτικών μέχρι και τη διανομή των αυτοκινήτων. Οι αντιπρόσωποι αυτοκινήτων τους οποίους εγώ άκουσα σε μία συνάντηση ιδιαίτερα επικοδομητική που είχαμε. Όλοι δεν είναι όλοι οι διανομείς οι οποίοι έχουν τα ίδια συμφέροντα. Έχουμε αντιπροσώπους, μεγάλα αντιπροσώπους, τα κράτη-μέλη με μεγάλη παρουσία στην αγορά αλλά έχουμε και πολλούς μικρούς οι οποίοι είναι πολύ πιο ευτυχείς με αυτά τα οποία προτείνουμε τώρα από ότι αυτό που ισχύει από το 2002 και μετά. Διότι ορισμένες, ορισμένα πράγματα ε, που δεν τα είχε ως στόχο νομοθέτης ε, τους εμπόδιζαν να σταθούν απέναντι στους μεγάλους. Έχουμε προβλέπουμε την προστασία, προβλέπουμε εξαιρέσεις. Όταν δηλαδή βλέπουμε εμείς ότι κάποιος πλήτεται και υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Μπορούμε εμείς με, τον ειδικό, με τις ειδικές ρυθμίσεις για τα αυτοκίνητα ή με κάθετες ρυθμίσεις να δίνουμε εξαιρέσεις. θεωρούμε ότι με τον τωρινό κανονισμό τα πράγματα θα διορθωθούν, όχι γιατί γίναμε πιο έξυπνοι μετά από 8 χρόνια, απλώς γιατί μεσολαβεί η εμπειρία που μας διδάσκει πολλά. Έχουμε το ψήφισμα για αυτό το σημείο και θα ψηφιστεί αύριο. Επόμενο σημείο.